συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα να μπορώ να καλωσορίσω έναν φίλο μας εδώ στο Κοινοβούλιο, τον πρόεδρο της ε, Σλοβενίας, Μπόρουτ Παχόρ, πρώην Ευρωβουλευτής. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω. Συνάδελφοι, ε, σε μια πρώτη συζήτηση που είχαμε τον Μπορούτ Παχόρ, ε, θέσαμε το ερώτημα, ο Τόμας Σίλβες, η Χέλε Τόρνινγκ Σμιτ, ο Ιώσεφ Μούσκατ, ο Μπορούτ Παχόρ, ο Τζόρζο Ναπολιτάνο, ο Έλιο Ντιρούπο, ο Φρανσουά Ολάντ, ο Ενρίκο Λέτα. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί. Είναι όλοι πρώην ευρωβουλευτές. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε. Βλέπετε τι μπορούμε να γίνουμε. Βλέπετε εδώ το παράδειγμα του Πρόεδρου της Σλοβενίας, κυρίες και κύριοι. Ε, χαίρομαι που μπορώ να δώσω το λόγο στον πρώην συνάδελφό μας. Ε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Господ председник, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, όπως μόλις είπε ο πρόεδρος, ο φίλος μου, ο Μάρτιν Σούλτς, ήμουν συναδελφός σας κατά την προηγούμενη θητεία. Ήμουν και προσωπικός φίλος κάποιων από σας. Να σας πω ότι μου λείπετε αρκετά συχνά. Και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο. Πολιτικά μου λείπετε. Όποτε συνειδητοποιώ ότι οι ευρωβουλευτές παίζουν, οι ευρωβουλευτές παίζουν ειδικό ρόλο στη δημιουργία της κοινή ευρωπαϊκής μας μοίρας. Πρόκειται για μια μοναδική θέση, η θέση του Ευρωβουλευτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαραίτητο, έχει ζωτική σημασία για τη διαμόρφωση της κοινή μοίρα μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Και ακριβώς γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απολύτως απαραίτητο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κυρίως θέμα σήμερα. Είναι ένα από τα θέματα ε, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά στους καιρούς μας. Και μαζί με σας που Έχετε απόψεις παρόμοιες με τις δικές μου. Ελπίζω να μπορέσω να συζητήσω το θέμα αυτό. Πρόκειται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό θέμα, θεωρητικό. Είναι θέμα ε, μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα είναι δύσκολο να καλυφθεί αργότερα στην σημερινή μου ομιλία θα ήθελα να κάνω ε, ένα νέο βήμα πολιτικό και νομικό για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ε, όχι παρά τις συνθήκες αλλά λόγω των συνθήκων έχουμε την κατάλληλη στιγμή για ε, ένα σημαντικό βήμα. Αυτή η στιγμή θα έρθει μετά τις ευρωεκλογές του χρόνου. Εύχομαι να έχουμε πάλι μια συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης και επιθυμία μου είναι οι εργασίες της συνέλευσης αυτής να ολοκληρωθούν με πολιτική πλειοψηφία ή ακόμα και συνένεση σχετικά με τις μελλοντικέ ανάγκες των ανθρώπων μας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ποιες είναι οι θέσεις σας. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς είναι αντίθετοι με τη θέση αυτή. Ξέρω ότι πολλοί έχουν αμφιβολίες σχετικά με την προσέγγιση αυτή και όλες αυτές οι αμφιβολίες είναι θεμητές και δημοκρατικές. Αυτό είναι ο λόγος άλλωστε που υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει για να έχουμε την ελευθερία να λαμβάνουμε αποφάσεις για το μέλλον πάνω στα πιο βασικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πνεύμα της, δικαιοσύνη, της δημοκρατίας. Κάποιοι είναι υπέρ, κάποιοι είναι κατά. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τη δική μου θέση. Τελικά, ο κόσμος ε, μάλλον θα θέλει να αποφασίσει πάνω στο θέμα αυτό με δημοψήφισμα σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος μέλος. Ε, κάτι που θα δώσει την πολιτική νομιμότητα σε μια τέτοια απόφαση και ο κόσμος έχει και δικαίωμα να απαιτήσει κάτι τέτοιο. Επιτρέψτε μου να δικαιολογήσω τη θέση μου και να σας προβάλλω δύο βασικά επιχειρήματα ε, σχετικά με το γιατί πιστεύω αυτά που πιστεύω. Ε, τα τελευταία 25 χρόνια είμαι πεπισμένος Ευρωπαίος. Πιστεύω στην ιδέα της Ευρώπης ως μια κοινότητα εθνών και κρατών. Και πιστεύω ότι παρά τις διαφορές μας ε, έχουμε περισσότερα κοινά τα οποία μας ενώνουν. Οι προηγούμενες εμπειρίες μας έχουν δείξει ότι η συνεργασία ε, αποτελεί εγγύηση για την ειρήνη και η ειρήνη οδηγεί σε ευημερία. Και άλλωστε το Νομπέλ Ειρήνης δείχνει ακριβώς αυτό. Ποτέ δεν εγκατέλειψα αυτές τις πεπιθήσεις μου. Αντιθέτως, η ευρωπαϊκή πεπιθήση μου έχει γίνει πιο ισχυρή. Μετά το, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Είδαμε σημαντικές προόδους, είδαμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας που αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα προόδου και σήμερα αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας σύντομα δεν θα αρκεί, δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του μέλλοντος. Δεν θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων που εκπροσωπούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική κρίση μας ε, έχει κάνει να σκεφτούμε τις ε, δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση, για περαιτέρω, ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλουμε να καλύψουμε το δημοκρατικό έλλειμμα και από το 2008 η οικονομική και κοινωνική κρίση έχει αποκαλύψει το συνολικό εύρος των προβλημάτων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Τα προβλήματα αυτά είναι πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής φύσης. Θα πρέπει ε, να ε, διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων μας ε, στο κοινό μέλος, μέλλον. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε 17-18 ε, διαφορετικές δημοσιονομικές πολιτικές. Κάτι τέτοιο είναι απλά αδύνατον. Βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να βρούνε προσωρινούς και μόνιμους τρόπους για κοινή δράση. Αλλά μακροπρόθεσμα κάτι τέτοιο δεν είναι αρκετά αξιόπιστη η βάση για τις νομικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θέλει να ενισχύσει και να αναπτύξει το ρόλο της ε, ως παράγοντας ε, στην διεθνή σκηνή. Το δεύτερο μου επιχείρημα είναι το εξής. Όπως ε, ανέφερε ο φίλος μου, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, έχω παίξει διάφορους ρόλους καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Οι περισσότεροι από εσά έχετε πίσω σας μακρά πολιτική σταδιοδρομία. Έχετε ποικίλε πολιτικές εμπειρίες, διαφορετικές αναφορές ο καθένας. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τις εμπειρίες που κερδίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ έχω και ε, εμπειρίες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι στις εποχές της κρίσης ήμουν, ε, ήμουν πρωθυπουργός και από το 2008 μέχρι το 2011 προσπαθήσαμε να βρούμε έδαφος να πατήσουμε και εξετάζαμε προσωρινές λύσεις ε, με αμφιλεγόμενη πολιτική βάση και χρειάστηκε να διορθώσουμε κάποιες αποφάσεις που είχαμε λάβει τότε επανειλημμένα. Ήμουν όμως εκεί και είδα από πρώτο χέρι ε, πώς αντιμετωπίστηκε η κρίση. Είδα πώς έπιασε η κρίση την Ευρώπη απροετοίμαστη. Και χωρίς ε, και δεν έχουμε κάποια θεσμικά όργανα τα οποία άλλοι έχουν στη διάθεσή τους ε, και γι' αυτό ο κόσμος κατηγορεί εμένα, εσάς, όλους, θεωρεί ότι είμαστε ανίκανοι. Θεωρεί ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να το κάνουμε αυτό. Και Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε στη διάθεσή μας τα κατάλληλα μέσα ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας. Ως Πρόεδρος της ε, Σλοβενίας μπορώ να σας πω ότι συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την κρίση Βλέπω όμως ότι υπάρχει μεγαλύτερη ενότητα ανάμεσα στις διάφορες δυνάμεις, ε, τις ε, κυβερνήσεις, ε, τα πολιτικά κόμματα. Μπορέσαμε να υιοθετήσουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες χρειάστηκαν μεγάλη οριμότητα και μπορώ να σας πω ότι η Σλοβενία θα ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και θα αποτελέσει και πάλι μια ιστορία επιτυχίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει όμως κάποια δυσπιστία απέναντι στα θεσμικά όργανα ε, και στο κράτος δικαίου. Έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα ε, βλέπουμε και στην Σλοβενία τα πρώτα δείγματα ευρωσκεπτικισμού. Από την άλλη όμως υπάρχει και ισχυρή πίστη, υπάρχει η γνώση ότι κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του ε, τα προβλήματα, μπορούμε όμως να το κάνουμε αυτό μαζί. Και αυτό ακριβώς είναι το πρωτεύον έργο μας αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε τις λύσεις θεωρώντας ότι στο μέλλον μπορεί να είναι πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Όχι, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ορμή που δόθηκε στην αρχή της χιλιετίας με την συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης. Πολλοί από εσά θα θυμούνται την εποχή αυτή. Θεωρήσαμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε τους στόχους της Λισαβόνας. Είπαμε ότι θα γίνουμε πιο ανταγωνιστική κοινωνία βασισμένη στη γνώση στον κόσμο. Ε, αποτύχαμε, αλλά μπορούμε να βγούμε από την παρούσα κρίση κάτι που θα δώσει νέα κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε επίσης εξυγίανση της οικονομίας, αλλά όλα αυτά θα σημάνουν ότι οι νέοι θα έχουν πάλι θέσεις απασχόλησης, οι νέοι θα έχουν την πίστη ότι θα ζουν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να τους εγγυηθεί μια αξιοπρεπή ζωή. Κύριε Πρόεδρε, η θέση μου όσον αφορά την ολοκλήρωση και εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, και τη διεύρυνση όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, ε, είναι εμπνευσμένη από ε, τη δουλειά μου εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη διεθνή πολιτική. Όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε μόνο με συνεργασία μεταξύ μας. Και αν θέλουμε ειρήνη διαρκείας, εάν θέλουμε περισσότερη ευημερία, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας. Το μήνυμά μου λοιπόν προς το Κοινοβούλιο σας και προς όλους στην Ευρώπη είναι ότι η κληρονομιά ειρήνης και ευημερίας που έχουμε μπορεί να προστατευτεί και να ε, αυξηθεί στο μέλλον, μόνο όμως με προϋπόθεση την πολιτική συνεργασία. Εάν διστάσουμε και δεν υιοθετήσουμε τις απαραίτητες αποφάσεις, κάτι τέτοιο θα διακυβεύσει την κληρονομιά αυτή. Το λέω αυτό ως πρόεδρος ενός μικρού ευρωπαϊκού κράτους. Μπορεί να θεωρούσατε πιο λογικό πρόεδρος μεγάλου κράτους να πει κάτι τέτοιο. Η Σλοβενία όμως έχει εμπειρίες από την κατάρρευση ε, ενός μεγαλύτερου ομοσπονδιακού κράτους και με τις εμπειρίες αυτές θα μπορούσα να συμβάλλω στους συλλογισμούς που αφορούν το μέλλον μας. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε λιγότερη κυριαρχία. Αλλά το αντίθετο συμβαίνει. Αυτή η μεταφορά αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της διαφορετικότητας σε κάθε κράτους, ε, των ιδιαιτεροτήτων ε, του κάθε κράτους. Ε, εάν δεν συνεργαστούμε, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς τη σύγχρονη ζωής. Και γι' αυτό είμαι ισχυρός υπέρμαχος της ε, περαιτέρω εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω την επιθυμία οι νέοι να μας στηρίξουν σε αυτές ε, τις φιλοδοξίες μας. Αλλά το 1 τέταρτο των νέων μας είναι άνεργοι. πολλοί από εμά μιλούμε για τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης χωρίς να ε, εξηγούμε στους νέους ότι αυτό θα ε, αποτελέσει, αυτό θα δημιουργήσει τις ε, συνθήκες ώστε να μπορούμε να ενεργήσουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να προοδεύσουμε στην επιστήμη και τεχνολογία, ότι αυτό θα μας κάνει αντιγωνιστικούς απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείε τη Βραζιλία και την Κίνα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους μας να καταλάβουν την έννοια της ε, περαιτέρω ε, ολοκλήρωσης. Ε, θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλα αυτά θα αυξήσουν τη δική τους ευημερία και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να καταβάλουμε προσπάθειες για κάτι τέτοιο. Το μέλλον μας εξαρτάται από τις προσπάθειες αυτές. Επιτρέψτε μου λοιπόν να δράξω την ευκαιρία να καλέσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα επιτρέψει στους νέους να βρουν αύριο θέσεις εργασίας. Είτε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ή μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους. Και εσείς, οι Ευρωβουλευτές, θα παίξετε σημαντικό ρόλο σε κάτι τέτοιο. Διότι θα συμμετέχετε και κατά την σύνοψη της συμφωνίας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για το διάστημα 2014-2020. Παρεπιπτόντως ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει παρεξήγηση. Όποτε μιλώ για τις ΗΠΑ Πολιτείες ε, της Ευρώπης ε, δεν έχω κατά νου το χωνευτήρι το αμερικανικό μοντέλο εμείς ε, θέλουμε να έχουμε ποικιλομορφία, διαφορετικότητα. Για να λειτουργήσει αυτή όμως υπέρ ημών, θα πρέπει να βρούμε μια νέα σχέση ανάμεσα στο σεβασμό της διαφορετικότητας και την ενθάρρυνση της ενότητας. Να είμαι απόλυτα σαφής. Και ξέρω ότι δεν συμφωνείτε όλοι μαζί μου, αλλά εάν είμαστε υπέρ μιας ισχυρής Ευρώπης, Και αν πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσουμε τις ιδέες μας, τελικά θα ε, υπερισχύσουν οι ευρωσκεπτικιστές και μπορεί να είναι μια βραχυπρόθεσμη νίκη για αυτούς, αλλά θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες ε, μια τέτοια αποτυχία από τη δική μας πλευρά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις, ε, την ευγνωμοσύνη μου απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, όσον αφορά την δημοκρατική λήψη αποφάσεων, ε, έχετε πολύ σημαντικό ιστορικό. Ξέρω ότι πολύ συχνά το κοινό δεν γνωρίζει αρκετά το ρόλο σας. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας ζητήσω να δεχτείτε την ευγνωμοσύνη μου και την ευγνωμοσύνη των πολιτών που εκπροσωπώ για τη δουλειά σας, για τις προσπάθειές σας προς όφελος των πολιτών μας. Προσβλέπω με πίστη στο κοινό μας μέλλον και πιστεύω ότι το Νόμπελ Ειρηνή δεν ήταν τόσο πολύ ε, αμοιβή, ήταν πιο πολύ προειδοποίηση ότι ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ειρήνη. Κάθε μέρα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να την πετύχουμε. Κάτι τέτοιο θα είναι η μόνη σταθερή βάση για την ευημερία των πολιτών μας και είμαι πεπισμένος ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μπορούμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ενθαρρυντική σας αυτή ομιλία. Πιστεύω ότι είναι μια ομιλία που θα οδηγήσει σε συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε στο Σύνταγμα της Ευρώπης, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνο όλους τους συναδέρφους μας. Ε, το ξέρετε αυτό. Η ενθάρρυνση για τις δικές μας εργασίες, κύριε Πρόεδρε, είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ε, πρώτη φορά ένας αρχηγός ε, κράτους ε, έχει ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για τις εργασίες του. Είναι και λογικό αυτό όμως, διότι κάποιος που τόσα χρόνια εργάστηκε ως Ευρωβουλευτής εδώ γνωρίζει ότι ότι, ε, ότι μια νομοθετική συνέλευση ε, με τόσα μέλη αποτελεί μοναδικό μέρος και σας ευχαριστούμε που μας ε, ενθαρρύνατε στις εργασίες μας. Κύριε Παχόρ, σας ευχαριστώ θερμά.